Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο βήμα στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα σχέδιο πίνακα αποτελεσμάτων για την επιτήρηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την κυρία Μπόλς, συντάκτη της προφορικής ερώτησης. You have the floor, Mrs. Um, Σας ευχαριστώ. Είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω να προχωρήσω. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έδωσε στη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον χρόνο να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με το scoreboard, το πίνακα βαθμολογήσεως και ε, να συζητήσει πριν υιοθετήσει το σχέδιο του πίνακα βαθμολόγηση των επιδόσεων μετά από διαβούλευση διαβούλευση. Ε, ναι. Υπήρξε μια πολύ ε, σαφή συζήτηση με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε το αποτέλεσμα και σχετικά με ε, ε, το πακέτο των έξι οδηγιών και παρόλο που τα τελικά μέτρα ακόμη είναι υπό εξέταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι ήταν πολύ σημαντικό να καθορίσει ανώτατα επίπεδα όποτε ήταν αναγκαίο και στο σχέδιο αυτό δεν αντικατοπτρίζεται για πολλούς από τους δείκτες βεβαίως δεν είναι πάντοτε προφανές να μπορεί κανείς να καθορίζει τα επίπεδα και τα όρια αλλά ε, πρέπει να εξηγήσουμε γιατί αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατόν και θα θέλαμε να ακούσουμε τα σχόλια της Επιτροπής επί του θέματος. Όσον αφορά τα πλεονάσματα επίσης χρειάζονται επεξήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι είπαν ότι όταν υπάρχουν χώρες με πλεονάσματα ή ελλείμματα στις τρέχουσες συναλλαγές θα πρέπει να προβλέπονται και οι αντιδράσεις και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την διόρθωση. Όλα αυτά έχουν σχέση με τις ε, ε, σχέσεις μεταξύ μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται στην οικονομική διακυβέρνηση χωρίς να μας δίνει τις αναφορές τις οποίες κάνει και οι οποία είναι αναγκαίες για να μπορέσει κανείς να καταλάβει τη μεθοδολογία. Ένας από τους στόχους της δημοσιονομικής ε, του δημοσιονομικού συντονισμού επίσης πρέπει να εξηγηθεί για να καταλάβουμε πώς θα λειτουργήσει ο πίνακας αυτός βαθμολόγησης και αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι το τέλος του 2012 θα υπάρξουν νέα κατόφλια σχετικά με τους δείκτες του οικονομικού τομέα. Εδώ αυτό έχει σχέση με ε, τους δείκτες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων. Ίσως είναι ένας τομέας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να περιληφθεί το ε, τον ε, μακροοικονομικό πίνακα βαθμολόγησης διότι βλέπουμε ότι στο άρθρο 4 ε, οι προτάσεις που κάναμε δεν έχουν ληφθεί υπόψη και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα συνυπολογιστούν στην αξιολόγηση του πίνακα κατά τρόπον ώστε να λάβουμε υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως ο ρόλος της ενεργείας και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό τον πίνακα βαθμολόγησης για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ρωτούμε λοιπόν πώς θα αξιολογούνται οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλα πλεονάσματα ή ελλείμματα εις ε, τον, ο, ετή, ετήσια έκθεση της προειδοποίησης ε, για τα προβλήματα. Επίσης ε, πόσο θα ερμηνεύεται οικονομικά ο πίνακας αυτός και τέλος σχετικά με τις αναφορές στη βιβλιογραφία και στη μεθοδολογία θα ήθελα να πω ότι μία ε, διάφανη εφαρμογή αυτού του συστήματος χρειάζεται για όλο το σύστημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας εξασφαλίσει ότι η λειτουργία του μέσου αυτού θα μπορούν να είναι προς όφελος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί μίας βάσεως ισότητος και σας ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνηση το λεγόμενο εξαπλό πακέτο, τέθηκε σε ισχύ χθε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εντατικοποιήσουμε τη χρήση και την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών. Σε δημοσιονομικό πεδίο έχει υπάρξει νομίζω πρόεδρος, σε μακροοικονομικό επίπεδο θα πρέπει να γίνουν και εκεί κινήσεις. Η πρότασή σας λοιπόν, κυρία Μπάουλς, για την βελτίωση του πίνακα επιδόσεων για τις μακροοικονομικές ελλείψεις ισορροπιών ε, είναι κάτι το θετικό. Σας ευχαριστώ για την προφορική σας ερώτηση που είναι ουσιαστικά εννέα ερωτήσεις προς τις οποίες θα προσπαθήσω στα δύο λεπτά που έχω στη διάθεσή μου και επτά δευτερόλεπτα να απαντήσω. Μετά από την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο και έχοντας πλέον τις απόψεις του Συμβουλίου από το μήνα Νοέμβριο, όπως επίσης και του Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνων από το Νοέμβριο, μπορούμε νομίζω να περάσουμε στην τελική εφαρμογή του πίνακα επιδόσεων χωρίς καμία καθυστέρηση και με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές. Ο τελικός αυτός πίνακας θα γίνει τμήμα του μηχανισμού έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου. Θα συζητηθεί και στο ΕΚΟΦΗΝ και στο Eurogroup ε, τον Φεβρουάριο τα λάβουμε υπόψη μας στις συζητήσεις και θα ξεκινήσουμε σε βάθος ελέγχους των μέτρων για τα κράτη-μέλη όπου χρειάζεται να υπάρξουν ακριβώς τα μέτρα αυτά και για τον μακροοικονομικό τομέα και για συστάσεις οι οποίες θα πρέπει να απευθυνθούν σε ορισμένα κράτη-μέλη αν αυτό είναι απαραίτητο. Εδώ υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην δημοσιονομική εποπτεία από τη μία την μακροοικονομική ε, από την άλλη. Και οι δύο θα έλεγα είναι προληπτικού τύπου, αλλά η εποπτεία η μακροοικονομική είναι φυσικά πιο μακροοικονομική από ότι η δημοσιονομική. Και γι' αυτό ακριβώς προαπαιτείται αν θέλετε η δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό το είδαμε και στην περίπτωση της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και οι δύο αυτές χώρες τα δημοσιονομικά τους πριν την κρίση πήγαιναν καλά αλλά αυτή τη στιγμή ξέσπασε η κρίση με όλη της την δύναμη και την ορμή αντιμετώπισαν πάρα πολύ σοβαρές μακροοικονομικές ανισότητες οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν σε δημοσιονομικά προβλήματα που προκάλεσαν ύφεση στην πραγματική οικονομία και σημαντικά κοινωνικά προβλήματα πλέον με ανθρώπινες και κοινωνικές σημαντικές συνέπειες. Η δημοσιονομική εποπτεία είναι θα έλεγα κάτι το ποσοτικό, το αριθμητικό, αλλά η μακροοικονομική εποπτεία είναι κάτι το οποίο απαιτεί θα έλεγα κάπως πιο θεωρητικές ε, προσπάθειες κατανόησης και πρόβλεψης. Όταν προτείνεται μια χώρα για μελέτη εις βάθος, αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα αυτή θα αντιμετωπίσει άμεσα μια κρίση. Αντίθετα σημαίνει ότι για τις συγκεκριμένες αυτές χώρες υπάρχει ένας κίνδυνος υπερβολικών προβλημάτων που αν επιβεβαιωθούν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Με άλλα λόγια, στην ουσία έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για προληπτική δράση η οποία θα έχει διορθωτικές επιπτώσεις επί αυτών των μακροοικονομικών ανισοτήτων ή ελλείψεων ε, ισορροπιών. Τώρα για την δίκαιη εφαρμογή ε, των προτάσεων αυτών για όλες τις χώρες. Η αξιολόγηση ε, θα έλεγα των συστημάτων τρεχουσών πληρωμών για όλες τις χώρες είναι κάτι το οποίο είναι αναπόστατο τμήμα του συστήματος και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μένει στη δήλωση που είχε κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 28η Σεπτεμβρίου. Τότε είχαμε πει ότι η εποπτεία η μακροοικονομική καλύπτει τις χώρες οι οποίες έχουν ελλείμματα και ε, φύση ε, μπορεί να υπάρχουν και διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ανάγκη και το κατεπήγοντα χαρακτήρα των διορθωτικών δράσεων που θα πρέπει να αναλυφθούν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη αγαπητά μέλη, να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι και οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 27 χώρες θα περάσουν μέσα από τη διαδικασία εποπτείας και νομίζω ότι από τα ευρήματα των μελετών αυτών θα ωφεληθούν και 27 χώρες προς το κοινό καλό. Είμαι βέβαιος ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο θα θελήσει να πάρει μέρος στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Εμείς από πλευράς μας θέλουμε και θα εμπλέξουμε κάθε μία χώρα ξεχωριστά της Ευρωπαϊκής Ένωση στη διαδικασία. Ο κανονισμός αυτός θα εφαρμοστεί σε όλους και για όλους προς όφελον κάθε κράτους μέλους του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κάτι το οποίο ξεχνάμε μερικές φορές όταν ε, μπλεκόμεθα σε πάρα πολύ ζωηρές συζητήσεις. Συνάδελφοι, τώρα θα πάρουν το λόγο μιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Θα σα παρακαλέσω να σεβαστείτε τον χρόνο, διότι πρέπει να φτάσουμε στι ψηφοφορίε. Έχουμε την ε, απονομή βραβείο Ζαχάροφ και θα στερώ τη δυνατότητα ομιλία όταν ξεπερνάτε τον χρόνο που έχει ήδη προβλεφθεί. Ξεκινάμε για την ε, ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ο κύριο Ντόρφμαν, για δύο λεπτά ακριβώ. Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, έχουμε συζητήσει πολύ εδώ για την ε, οικονομική διακυβέρνηση ε, και το σύνολο των έξι οδηγιών, το Six Pack και ε, χθε επιβεβαιώθηκαν οπότε η μακροοικονομική επιτήρηση πρέπει να φέρνει στο επίκεντρο των συζητήσεων των πίνικων ε, επιδόσεων και πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να επεξεργαστεί τον πίνακα επιδόσεων πράγμα το οποίο έχει κάνει, το έχουμε μπροστά μας αλλά δεν είναι ακόμη πλήρως ικανοποιητικό. Στην πολιτική μας συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε επικεντρωθεί στην αξιολόγηση του πακέτου των έξω οδηγιών αλλά διαπιστώνουμε ότι ακόμη και αν δεν ευσταθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μία εσωτερική αγορά η οποία κινείται διμερός και αποβλέπει στο να εξέγει ε, στη σημερινή εποχή θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά αγορά. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς να πει ε, να προσάπτει σε ένα κράτος ότι δεν κάνει το καθήκον του εάν οι άλλοι δεν είναι άψογοι. Θα αναπτυχθεί αυτός ο πίνακας επιδόσεων, θα χρειαστεί χρόνο, άλλα στοιχεία θα συμπεριληφθούν, οριακές τιμές θα πρέπει να βελτιωθούν, γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προβλέψει να ε, επιτηρεί αυτή την εξέλιξη στηρίξει και να την αξιολογήσει και με την συνδρομή σας κύριε Επίτροπε θα το πράξουμε. Το ΕΛΚ έχει αξιολογήσει σαν θετικό το έγγραφο που έχει ε, υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. κυρία Ποδηματά. Ε, δύο λεπτά κυρία Ποδηματά. Πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το χθεσινό φίλο του, η Financial Times, δημοσίευσαν ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο γιατί η συμφωνία της 8 η δεκεμβρίου για τη δημοσιονομική ένωση θα αποτύχει με μια σειρά απολογικά και αυτονόητα θα έλεγα επιχειρήματα πολλά από τα οποία έχουν υποστηριχθεί και υποστηρίζονται εδώ και καιρό από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και ιδιαίτερα από την ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών η εφημερίδα επισημαίνει ότι είναι αντιπαραγωγική η μονομερής αιμονή στη δημοσιονομική πειθαρχία γιατί όπω σημειώνει η ορθή δημοσιονομική συμπεριφορά και πάλι μπορεί να συνδέεται με τεράστιε ανισορροπίε και με οικονομική αναποτελεσματικότητα και ε, επικαλούμενο ο αρθρογράφο το παράδειγμα τη Γερμανία, η οποία όπω γνωρίζετε πέρσι είχε πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τη τάξη του 5,7% του αεπ μεγαλύτερο και από αυτό τη ε, Κίνα. Ε, ο αρθρογράφος επιλέξει σημειώνει ότι το σύμφωνο ε, της δημοσιονομικής ένωσης θα αποτύχει γιατί δεν προσφέρει καμία απολύτως εξήγηση για το πώς ακριβώς αυτό το πλεόνασμα το γερμανικό θα ανακυκλωθεί όταν ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες χώρες του νότου αλλά όχι μόνο παραμένουν θρησκευτικά προσιλωμένες στην αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και ορθοδοξία γι' αυτό κύριε επίτροπε κύριε αντιπρόεδρε της επιτροπής θεωρούμε την ε, αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών όχι μια αποσπασματική συμφωνία αλλά μια βασική αρχή η οποία πέρα από το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να συνδεθεί άρρηκτα και με το νέο δημοσιονομικό ε, σύμφωνο τη δημοσιονομική ένωση όπως ε, αποκλήθηκε. θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι κομβικό σημείο για την επίτευξη συμφωνίας στους δύο κανονισμούς ήταν η σαφής δήλωση δική σας της ευρωπαϊκής επιτροπής ότι η διαδικασία θα αφορά τόσο σε κράτη μέλη με πλεονάσματα όσο και σε κράτη μέλη ε, με ελλείμματα καθώς επίσης και σε ανώτατα και κατώτατα όρια ώστε να υπάρχει συμμετρία. και αυτό δεν είναι μια δογματική αρχή είναι μια προϋπόθεση για να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία θα έχει πραγματική οικονομική σύγκληση με συγχωρείτε σας το επεσήμανα ήδη δεν έχουμε χρόνο. Ε, θα προχωρήσουμε στην ομάδα των φιλελευθέρων. ο κύριος χάγκλουντ για δύο λεπτά ακριβώς δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η οικονομική κρίση απέδειξε ότι και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες μπορούν να διακυβεύσουν την ευρωπαϊκή οικονομία παρά υγιή, σχετικά υγιή οικονομικά. Οπότε όσοι θεωρούσαν ότι τέτοιες επιδόσεις δεν είναι απαραίτητες, σφάλουν. Νομίζω είναι μεγάλη προσπάθεια για τη μακροοικονομική επιτήρηση και νομίζω ότι τα αποτελέσματα γενικώ είναι πολύ θετικά. Ε, βλέπουμε τώρα τα πρακτικά αποτελέσματα αυτή τη λύση. Είμαι προσωπικά πεπισμένο και η ομάδα μου το ίδιο ε, για το θετικό έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αρχική πρόταση. Πάντω είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι αυτό είναι το σημείο φετηρία τη μακροοικονομική επιτήρηση. Και δεν θα πρέπει από τώρα να διωγγώσουμε το ρόλο της στην ε, συνολική διαδικασία. Ο πίνακας επιδόσεων είναι μηχανισμός προειδοποίησης και χρειαζόμαστε και εξονυχιστικές μελέτες για να δούμε που υπάρχουν τα προβλήματα και που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η διοκτησία αυτού του σχεδίου δεν θα πρέπει να ανήκει η κυριότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια αυτό διεκδικεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι οι κύριοι, να έχουν την κυριότητα, την ιδιοκτησία αυτού του σχεδίου και να χαίρουν τη ε, συνδρομή και τη συμβουλή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι την κυριότητα θα πρέπει να την κρατήσουν τα κράτη-μέλη. Ε, είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε αποτελέσματα και να είναι λειτουργική αυτή η διαδικασία. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι πρέπει όλοι είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι το εξαπλό θετικό πακέτο που τέθηκε σε ισχύ αυτή την εβδομάδα ήταν σημαντικό βήμα ε, προς το δρόμο της διεξόδου από την κρίση. Και όλοι εκφράσαμε την ικανοποίηση μα γι' αυτό και για το γεγονό ότι τόσο σοβαρά έλαβε υπόψη το έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον χρόνο. Ο κύριο Λάμπερτ για 1,5 λεπτό, παρακαλώ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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, στις επιχειρήσεις όπως και στη ζωή η βάση όλων είναι η εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι ε, εσείς προδώσατε αυτή την εμπιστοσύνη σε τρία σημεία. Πρώτον, διότι σας είπαμε ότι το Κοινοβούλιο δεν θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα να συναποφασίσει τους δείκτες ε, βάσει ενός φίλου πορείας ότι θα μας θα σας παρακολουθούσαμε εκ το σύνεγγις ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Συμβούλιο και δεν θέλω να ξέρω με ποιες λεπτομέρειες ε, κατέληξαν στο Κοινοβούλιο και μας είπαν έχουμε ετοιμάσει κάτι, είσαστε ικανοποιημένοι. Δεν είναι σωστό. Ε, διαλέξατε τον, ε, τον συνεργάτη σας και δεν νομίζω ότι επιλέξατε σωστά. Διότι αυτά δεν είναι όλα όλα τα ίδια. Όταν μας λέγουν ότι οι χώρες που έχουν πλεόνασμα δεν θα τιμωρούνται, είναι να θεωρεί κανείς ότι τα πλεονάσματα δεν είναι επικίνδυνα, ενώ πιστεύω ότι τα υπερβολικά πλεονάσματα είναι εξίσου επικίνδυνα όσο και ε, τα ε, υπερβολικά ελλείμματα. Τέλος, η ε, μισθή που είναι η η έλλειψη ε, της ε, ανταγωνιστικότητας όπως είπατε δεν μπορεί να μας καταστήσει εκείνα όπου δεν θα έχουμε ποτέ τόσο χαμηλούς μισθούς. Από χθες, αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε έναν νέο μηχανισμό επιτήρησης ε, που λειτουργεί και θα ήθελα ε, να ξέρω ποια είναι τα ε, επικίνδυνα θέματα που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Κοινότης διότι εδώ θεωρούμε ότι 3% υπέρβαση του ελλείμματος είναι επικίνδυνο αλλά η μείωση των μισθών δεν είναι τι θα γίνει με τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη διότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αυξηθεί η οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, ο πίνακας επιδόσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι διότι οι στατιστικές δεν επιλύουν τα πράγματα εφόσον ο δείκτης αυτός τιμωρεί τις χώρες οι οποίες έχουν αποκλειστεί αποκλίνει και θα πρέπει να αποσυρθεί το σύστημα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα συζητάμε περί κανόνων και ρυθμίσεων, κάτι το οποίο θα αλλάξει άρδιν μετά από τις αποφάσεις της περασμένης εβδομάδας που έβαλαν η Γαλλική και Βρισκόμαστε ενώπιον αυτής της δύσκολης επιλογής, αν και στο παρελθόν υπήρχαν διάφορες ρυθμίσεις για την πρόληψη ανισορροπίων μέσω του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο υπογράφηκε το 1997. Αυτή η συμφωνία όμως κατέστη ε, σκουπιδό χαρτό διότι η Γαλλία και η Γερμανία τον τροποποίησαν άρδιν. Εγώ δεν είμαι διόλου ενθουσιώδης ε, οι Βρυξέλλες ε, να είναι ο άγνητος φύλακας και να μας επιβάλλει κάποιες ε, διευθετήσεις. Αλλά νομίζω ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να την χάνουν της ίσης αντιμετώπισης. Συμπεριλαμβάνουμε και των κρατών που σήμερα μας κάνουν το δάσκαλο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ισότιμη αξιοπρέπεια όλων των κρατών και να γίνονται σεβαστοί, σεβαστοί από όλους. Στη διαδικασία Catch the Eye, ε, παρακαλώ θα πάρουν το λόγο πέντε συνάδελφοι ε, έχουν ζητήσει το λόγο παραπάνω, αλλά θα κρατήσετε το ένα λεπτό σας παρακαλώ. Ο κύριος Γκούτας. Κούτας, ο κύριος Κούτας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε το ζήτημα των, ε, της επιθύρησης των μακροοικονομικών ανισορροπιών νομίζω ότι είναι σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη της σύγκλησης ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Εδώ θα πρέπει να συμπεριληφθεί η ανάλυση όλων αυτών των ε, ισορροπιών, ανισορροπιών που υπάρχουν και να ε, προλαμβάνεται το έλλειμμα, το υπερβολικό, όπως δυστυχώς συνέβη μέχρι τώρα. Ε, θα πρέπει λοιπόν η επιτήρηση αυτήν των μακροοικονομικών ισορροπιών να μην μπορέσει να παρεμποδίσει μια πραγματική δημοσιονομική πολιτική ευρωπαϊκή. Τα μέτρα λοιπόν αυτά δεν ε, προσφέρουν τίποτα άλλο από το να καθιστούν πιο άθροστες τις κοινωνίες και να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην πράσινη τεχνολογία, στις υποδομές, έτσι ώστε να ε, βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση στην Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με το, μέτρο αυτό του υποθέμενου οικονομικού συντονισμού τελικά επιμένουμε στην εμβάθυνση της καπιταλιστικής ολοκλήρωσης με τα γνωστά αποτελέσματα. Αύξηση της απασχόλησης, επιδείνωση της φτώχειας και των κοινωνικών uh, ανισοτήτων. Και αυτό αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διαδικασία δείχνει αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι να ε, ενισχύσουμε τη δινή κατάσταση των εργαζομένων αυξάνοντας ε, το μισθολογικό κόστος και ε, διευκολύνοντας τη συσσόρευση κεφαλαίου και επιδεινώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες. Ταυτόχρονα με την πρόταση αυτή θα διακυβεύσουμε τα συμφέροντα των χωρών που έχουν τις ασθενέστερες οικονομίες επιβάλλοντάς τους ε, ε, χειροπέδες ουσιαστικά και ε, πλήττοντάς τους με κυρώσεις που θα οδηγήσουν ακόμη πιο δίνη κατάσταση. Αυτή είναι μια απαράδεκτη επέμβαση και περιφρόνηση των στοιχειωδών αρχών της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Το λόγο ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι ενάντιος εις τις ανισορροπίες και εις ε, τα πλεονέασματα ε, διότι σωστό είναι να υπάρξουν κυρώσει, κυρώσεις αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις και για τα πλεονάσματα και για τα ελλείμματα και ε, βεβαίως εάν είχαν χρησιμοποιηθεί αυτές οι ε, δυνατότητε ε, θα είχε καταρρεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπάρξει ε, μία χωριστή ζώνη μεταξύ της Γερμανίας, Ολλανδίας, της Γερμανίας και να αφήσουμε τις άλλες χώρες να μπορέσουν να υποτιμήσουν τα νόμισμά τους. I can only hope that the unsustainable nature of the path chosen has become as evident as it is ultimately self-defeating for the whole Union. Με το ίδιο νόμισμα χωρίς ε, δυνατότητα ε, υποτίμησης, οι περιφερειακές ε, χώρες περιορίζονται σε ανάστροφο πληθωρισμό, ενώ οι μισθοί συμπιέζονται. Τα προβλήματά μας δεν λύνονται εύκολα. Εμείς στα άκρα της Ευρωζώνης έχουμε υποστεί σημαντικά πλήγματα και προβλήματα και στο μέλλον μας υπόσχονται ακόμα περισσότερα από τις πολιτικές, ε, λόγω των πολιτικών εξελίσεων. Πού είναι η αλληλεγγύη. Ε, με τα ε, ε, υψηλά επιτόκια δεν μπορούμε να επιζήσουμε. Χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση που να βοηθάει όλους τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Πολύ. Και ο κύριος Πάσκα, τελευταίο παρεμβαίνων. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Súčasťou procedúry a prevencií náprave makroekonomických nerovnováh má byť aj mechanizmus Χρειάζεται ένας ε, μηχανισμός ε, προληπτικός ε, που θα ειδοποιεί σχετικά με ελλείμματα των κρατών μελών. Κατά αυτόν τον τρόπο θέλουμε να αξιολογήσουμε τις ανισορροπίες και γι' αυτό δημιουργείται αυτό το scoreboard για να μπορούμε να δίνουμε αποτελέσματα σχετικά με χώρες και οι αποφάσεις που βγαίνουν από την έκθεση αξιολόγησης είναι σημαντικές και θα πρέπει τα στοιχεία να είναι πραγματικά αντικειμενικά και ορθά. Τα στοιχεία θα πρέπει να εμφανίζονται στο scoreboard κατά τέτοιο τρόπο ώστε ε, να μην υπάρχει δυνατότητα δημιουργικής λογιστικής ή επηρεασμού των δεδομένων. Πίτροπος, ε, Mr. Commissioner, you have the floor. Dear colleagues, could you take... Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ τους συναδέλφους να καθίσουν με ησυχία. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ε, σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση και για την ε, υποστήριξη που εκφράσατε σε αυτόν τον ε, κανονισμό και στις δράσεις της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα της κυρίας Μπόλς. σε ό,τι αφορά το πίνακα βαθμολογία και το πού στηρίζεται. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε ένα επεξηγηματικό έγγραφο που θα εξηγεί το οικονομικό σκεπτικό ε, πίσω από τις επιλογές των δικτών που κάναμε συμπεριλαμβανομένων και αναφορών σε οικονομική τεκμηρίωση ε, εγώ αναλαμβάνω προσωπικά την ε, δέσμευση ε, ότι η Κομισιόν θα σας παράσχει αυτές τις πληροφορίες που αφορούν, όπως σας είπα, το οικονομικό σκεπτικό μας. Η κυρία Ποδηματά αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο μέσον βρετανικό δεν νομίζω ότι είναι θέσφατο τα λόγια της ε, ε, του συγκεκριμένου μέσου. Ε, στο ίδιο μέσο η Ευρωζώνη, σας υπενθυμίζω, είχε χαρακτηριστεί όχι ως μικρή ανοιχτή οικονομία, αλλά ορισμένοι σχολιαστές θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη κλειστή οικονομία. Όχι, δεν είναι μια μεγάλη κλειστή οικονομία. Αντιθέτως είναι μια μεγάλη ανοιχτή οικονομία. Ένα που εμπορεύεται ένα μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ με τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό έχει προφανείς συνέπειες στον, στη δόμηση του αναλυτικού μηχανισμού μας για τον έλεγχο των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η νομοθεσία ακριβώς αντικατοπτρίζει την ε, ευφυή συμμετρία σύμφωνα με την οποία η επιτήρηση καλύπτει και τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα αλλά υπογραμμίζει ότι υπάρχει, είναι πήγον να αντιμετωπίσουμε περισσότερο τα μεγάλα ελλείμματα και γι' αυτό πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πολιτικές μας α, απαντήσεις. Το άρθρο 3.2 αναφέρει η έκθεση ότι η αξιολόγηση των κρατών μελών που όταν δείχνει μεγάλα ελλείμματα μπορεί να διαφέρει από την αξιολόγηση των χωρών που έχουν σωρεύσει μεγάλα πλεονάσματα. Ε, νομίζω ότι ο θόρυβος ε, δείχνει ότι ε, δεν είναι δυνατό να συνεχίσουμε περισσότερη αναλυτική συζήτηση για αυτό το θέμα, οπότε προτείνω να συνεχίσουμε το διάλογο μας στην Επιτροπή ΕΚΟΝ σε λίγο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα μια πρόταση ψηφίσματο για το τέλο αυτή τη συζήτηση. Έληξε εδώ όμω η συζήτηση αυτή και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στι 11.30 το μεσημέρι. Σα ευχαριστώ πολύ.